Το επόμενο σημείο λοιπόν είναι η προφορική ερώτηση της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας σε σχέση με την ποιότητα των καυσίμων και ιδίως για... Α, λάθος διαβάζω, λάθος θέμα διαβάζω. a ver qué punto Ε, διορθώνω, διορθώνω, λέει ο πρόεδρος. Δεν ανέγνωσα το σωστό σημείο της μερισιάς διάταξης. Άλλο είναι το σημείο που έπεται. Και συγκεκριμένα είναι η έκθεση του κυρίου ΣΒΑΠ για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Το λόγο έχει ο εισηγητής, κύριος ΣΒΑΠ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Καταρχάς ε, να πω ότι και δεν το κάνω από απλή ευγένεια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που συνεργάστηκαν για το συμβιβασμό και για την οδηγία που συζητάμε ε, σήμερα. Την κυρία Γουόλης, τα μέλη της Επιτροπής Ζουρί, την κυρία Γκέπχαρτ, τον κύριο Ροσφόρ, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, τον κύριο Βίλαντ. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν ήταν πάντοτε απλή και γι' αυτό χρειάστηκαν και δύο χρόνια για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Είχαμε 2.000 τροπολογίες και θέλω να ευχαριστήσω όλου όσου συνεισέφεραν σε αυτό το αποτέλεσμα. Μπορεί να έχουμε διαφωνίε ή διαφορέ σε κάποια σημεία και θα τι ε, δείτε και στι συμβαστικέ προτάσει. Παρ' όλα αυτά, καταλήξαμε σε συμφωνία όλε οι πολιτικέ ομάδε για να προχωρήσουμε με την εσωτερική αγορά προ όφελο των επιχειρηματιών και των καταναλωτών. 20 χρόνια μετά την ενία αγορά και την θέσπιση, την ενία πράξη συγγνώμη και την ενία αγορά, διαπιστώνουμε ακόμα ότι δεν υπάρχει παρόλο τους κανονισμούς και οδηγίες καμία εναρμόνιση. Συχνά δικαίω, αλλά συχνά και αδίκως οι χώρες μέλη εκμεταλλεύονται κάθε περιθώριο που διαθέτουν. Τώρα πάμε να φτιάξουμε την μέση οδό που θα ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο ορισμένα θέματα ενιαίας αγοράς αλλά θα αφήνει και περιθώριο λήψη απόφασης σε χώρες μέλη. Μπορούμε να προχωρήσουμε αρκετά σημαντικά και μάλιστα υπερκομματικά. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίξαμε και σωστά κάναμε την θέση της Κομισιόν έχοντας βελτιώσει κιόλα την ίδια πρόταση αρκετά η, ώστε η προστασία του καταναλωτού να λάβει τη θέση που της αρμόζει μέσα στην οδηγία αυτή προβλέποντας δικαίωμα ανακλήσεως η ε, καταγγελία της ε, συμβάσεις από πλευρά καταναλωτού μέσα σε 14 ημέρες για οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συνάψει με ηλεκτρονικό τρόπο. Φροντίζουμε ώστε να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στις ε, συμβάσεις μέσω διαδικτύου και καταπολεμούμε έτσι κάθε είδους απάτη. Επιβάλλουμε και υποχρέωση ενημέρωσης για κάθε σύμβαση που γίνεται μέσω διαδικτύου σε ό,τι αφορά τις τιμές. Ωστόσο κάναμε την ε, οδηγία αυτή και εύχριστη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις φροντίζοντας ώστε να γίνουν οι προσφορές υπηρεσιών εύκαμπτες, να υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις για αυτές, να επιτρέπεται η, ε, σύναψη, ε, η διαφήμιση από το τηλέφωνο, να Επιτρέπουμε ωστόσο να έχουν οι καταναλωτές ξεκάθαρους όρους για την επιστροφή του προϊόντος εφόσον δεν συμφωνούν με αυτό. Και με ένα έντυπο το οποίο να επιτρέπει την επιστροφή του εμπορεύματος πανευρωπαϊκά θα παρακολουθήσουμε την ε, εξέλιξη του δικαίου στον τόσο σημαντικό αυτό τομέα. Θα το κάνουμε πολύ λιγότερο περίπλοκο από ό,τι στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να συνεννοηθεί ευκολότερα με το Συμβουλίο, διότι ενιαία αγορά χρειάζεται ενιαίους κανόνες. Τα είδαμε αυτά τα πράγματα πολύ καθαρά στην κρίση του ευρώ. Δεν αρκεί να τάσεται κανείς υπέρ κοινών αρχών, και να αφήνει κάθε διακριτική ευχέρεια στις χώρες μέλη, πρέπει οι κοινέ αρχές να εφαρμόζονται και με κοινού κανόνες. Και αυτό εξασφαλίζουμε. Για τους καταναλωτές στην οδηγία αυτή, ακόμα καλύτερα διότι θα γνωρίζουν τα δικαιώματά τους εφόσον αυτά είναι ενία και θα μπορούν να αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν τα σέβονται. Το ίδιο θα υπάρξει ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τότε θα μπορέσει πραγματικά να ανθίσει αυτή η πολιτισμική ποικιλία που τόσο συχνά επικαλούμαστε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξενόματος του Συμβουλίου έχει το λόγο κυρία Γκέρι. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κύριε Σφάμπ, Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική πρόταση και ανταποκρινόμεθα σαν Συμβούλιο με πολύ ενδιαφέρον και σαν Προεδρία. Ήδη από τον προηγούμενο χρόνο το Συμβούλιο κατέληξε στην προκαταρκτική του θέση τις γενικές θέσεις στις 24 Ιανουαρίου του 2011. Η συμφωνία πήρε δύο χρόνια. Δύο χρόνια προσπαθήσαμε να δούμε ποια θα ήταν η καλύτερη ισορροπία για να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα των καταναλωτών και το περιβάλλον και πώς θα μπορούσαμε να εναρμονίσουμε τους, ε, τους τρόπους προστασίας των καταναλωτών. 60 συναντήσεις χρειάστηκαν στο Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε μια ενισχυμένη πλειοψηφία. Δεν υπήρξε συμφωνία στα κεφάλαια 4 και 5 σχετικά με την πώληση προϊόντων με συμβόλαια τα οποία δεν ήταν ισχυρά. Και γι' αυτό αναγκαστήκαμε στο Συμβούλιο να διαγράψουμε αυτά τα δύο κεφάλαια και να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα κομμάτια των συμβάσεων που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η στάση αυτή υποστηρίχθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ήδη το εναπομείναν κείμενο του Συμβουλίου προσέφερε προστιθέμενη αξία σε σχέση με την βελτίωση των συμβολέων συμβάσεων αυτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερο και γι' αυτό η ψηφοφορία την οποία θα τελέσετε αύριο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εάν η Ολομέλεια αποφασίσει να παραπέμψει εκ νέου το θέμα προς την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, σαν Ουγγρική Προεδρία θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να πετύχουμε τον συγκεκριμένο στόχο και πάρα πολλά βέβαια θα εξαρτηθούν από τις τροπολογίες οι οποίες θα κατατεθούν από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως σας έχω ήδη πει υπάρχει πολύ σημαντική διαφορά σχετικά με το περιεχόμενο ιδιαίτερα των κεφαλαίων πάντα 4 και 5 που είναι σε εκκρεμότητα. Συνθήκες πώλησης προϊόντων, εγγυήσει των προϊόντων τα οποία πολλούνται και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να εναρμονιστούν όλα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σαν Προεδρία πιστεύουμε ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα πλέον να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο 1 και στο 3, όπου εκεί υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ε, ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο όπως το έχει ψηφίσει η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Ίνκος στις αρχές του μηνός Φεβρουαρίου και τα τέλη Ιανουαρίου οι άλλοι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, θα συνεργαστούμε και με εσά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε και με τις προτάσεις σας, να καταλήξουμε από κοινού κάπου και σας ευχαριστώ προκαταβολικά για την προσπάθεια την οποία κάνετε και εσείς και τα κράτη-μέλη βέβαια δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική κατάληξη αυτής της προσπάθειας, αλλά είμαι πεπισμένη ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία αυτή και να σημειώσουμε πρόοδο εκεί τουλάχιστον όπου πρόοδος μπορεί να σημειωθεί. Και ελπίζω έτσι να κατανοήσει ο Ευρωπαίος πολίτης ότι θα του έχουμε διασφαλίσει περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν δικαιώματα. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το λόγο έχει η Επίτροπος Ρέντινγκ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, του χρόνου εορτάζουμε την 20η επέτειο από την ίδρυση εσωτερική αγορά και θα πρέπει τη ενιαία αγορά, μάλλον. Και θα πρέπει η ενιαία αυτή αγορά να φέρνει ωφέλη. Ωφέλη στου καταναλωτέ αλλά και στι επιχειρήσει. Πάνω από δύο χρόνια ε, κράτησαν οι διαπραγματεύσει και αυτό έδειξε ότι από πολιτική πλευρά είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει συμφωνία ε, σε σχέση με το σύνολο τη οδηγία επί τη βάση των προτάσεων τη Κομισιόν και πολλοί από εσά σωστά δεν θέλετε να δείτε μείωση των επιπέδων της εθνικής προστασίας των καταναλωτών. Τώρα βρισκόμαστε πια στον τρίτο χρόνο της συζήτησης αυτού του νομοθετήματος και νομίζω ότι καιρό είναι πια οι συνομοθέτες να βρουν μια λύση. Και θέλω γι' αυτό ακριβώς ε, να ευχαριστήσω τους τη της Επιτροπής σας, ΣΦΑΠ, ε, αλλά και τους σκιώδεις συζητητέ για τη σκληρή τους δουλειά για την εξέβρεση ενός συμβιβασμού. Το Συμβούλιο αποφάσισε αρχές του έτους ε, για μια γενική προσέγγιση, δηλαδή να περιορίσει σημαντικά το εύρος της πρότασης και να στοχεύσει συγκεκριμένα στις ε, από απόσταση πωλήσει ε, και σε πωλήσει εκτός πρατηρίων στόχος είναι να βρούμε μια καλή ε, συνένεση και ο, νομίζω ότι ο συμβιβασμός ουσιαστικά βελτιώνει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς αλλά παρέχει και προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές. Αυτός είναι ο στόχος. Ξέρω ότι η συστροπολογία σας επιδιώκεται περαιτέρω βελτιώσεις. Και βλέπω επίσης πολλές λογικές υποδείξεις για περαιτέρω αυξήσεις προστασίας των καταναλωτών. Και όπως προείπα, τα δικαιώματα των καταναλωτών, η σχετική οδηγία δηλαδή, θα πρέπει ακριβώ αυτό να αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών για να αξίζει το όνομα που φέρει. Θέλω να σα δώσω κάποια ε, παραδείγματα. Θα μπορούσα να δεχθώ πολύ καλά την τροπολογία 122 που εξασφαλίζει ότι οι καταναλωτέ ε, δεν θα επιβαρύνονται αν στείλουν πίσω εμπορεύματα εάν αυτά αξίζουν πάνω από 40 ευρώ μετά την απόσυρσή του, Ούτε είμαι αντίθετη η περίοδο τη ε, της να επεκταθεί στον ένα χρόνο εάν δεν είχε ενημερωθεί για το σχετικό δικαίωμα ο καταναλωτή. Ε, πρόκειται για τροπολογία 116. Μπορώ επίση και την εναρμονισμένη λύση για την καταπολέμηση ε, των λεγόμενων Internet Cost Traps, αυτών των διαδικτυακών παγίδων στην τροπολογία 107 και παράγραφη 1α ε, και 1β Βέβαια δεν θα σας εκπλήξει το ότι εγώ δεν μπορώ να δεχθώ όλες τις τροπολογίες σας. Δεν μπορώ να δεχθώ όλες τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει και για παράδειγμα την τροπολογία 141 παρότι ο στόχος μου και εμένα είναι να υπηρετήσουμε την ενιαία αγορά. Θεωρώ πάντως ότι πηγαίνουμε λίγο μακριά αν οι εξαποστάσεως ε, πολιτές ε, πρέπει να ε, πληρούν κάποιες περαιτέρω προποθέσεις ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών ή πώληση προγραμμάτων σε τρίτες, σε άλλες χώρες. Πάντως εγώ βλέπω φως ε, στην άκρη του τούνελ. Είμαι πεπισμένη ότι μια ισορροπημένη και αποδεκτή συμβαστική λύση πλέον είναι κοντά και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας βοηθήσω να φτάσουμε σε αυτή τη λύση. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο εκ μέρους Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Αυτό λόγο η κυρία Γουόλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Από κοινού έχουμε κάνει μια μεγάλη διαδρομή και ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτό το κοινό ταξίδι και να καταλήξουμε στον προορισμό μας. Ευχαριστώ τον εισηγητή από πλευράς της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων Είδαμε στα τελευταία χρόνια τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω της ύπαρξης των διαφορετικών νομικών ενιών και αντιλήψεων σχετικά με τον τρόπο που θα λειτουργούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά. Έχει υπάρξει κάποια πρόοδος πάντως. Δυστυχώς όμως Ίσως έχουμε ξεπεράσει τα όρια, έτσι τουλάχιστον πιστεύουμε εμείς, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 5 ε, για τις ε, ρήτρε οι οποίες φύγουν τον καταναλωτή, ιδιαίτερα στον τομέα της διαφάνειας. Εκεί θα θέλαμε να υπάρξει περισσότερη πρόοδος και ελπίζω ότι το Συμβούλιο ίσως έχει κάνει ένα βήμα επιπλέον ή μάλλον πρέπει να κάνει ένα βήμα επιπλέον το οποίο πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη σημασία για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Συνεπώς λοιπόν έχουμε καλύψει μεγάλη απόσταση. Προστατεύουμε το κοινοτικό κεκτημένο σε σχέση με τα δίκαια του καταναλωτή. Δεν έχουμε συμφωνήσει σε όλα τα θέματα βέβαια, έχουμε κάνει όμως κάποια μικρά βήματα. Ελπίζω να συνεχίσουμε αυτά τα μικρά βήματα και ελπίζω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε κάπου. Ευχαριστώ κύριε Βόλης. Είναι εντός, ε, η κυρία Πιατικά είναι εντός της αιθούσης. Εκ μέρους λοιπόν ε, της Επιτροπής Οικονομικών και νοσματικών Υποθέσεων για δύο λεπτά έχετε το λόγο κυρία είναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για τη συνεργασία και ιδιαίτερα τον κύριο Σφαμ από την ΙΜΚΟ για τις ατέρμονες προσπάθειες και το συνεργατικό πνεύμα που επέδειξε με στόχο να περάσει αυτή η πρόταση, γιατί πράγματι η πρόταση της Κομισιόν ε, άφησε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Από την πλευρά τώρα της Επιτροπής ΕΚΟΝ, τρία θέματα θα ήθελα να θέσω. Πρώτον, είναι καλό που τα ψηφιακά αγαθά έχουν περιληφθεί στην πρόταση. Είναι καλό που υπάρχει ένα σαφές μήνυμα για την ανάπτυξη εναλλακτικών μηχανισμών επίλυση διαφορών στο μέλλον. Και αυτό αφήνει και κάποια ελπίδα για το μέλλον. Και συγκεκριμένα όταν μιλάμε για μικρά ή καινοτόμα χρηματικονικά προϊόντα, αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται είτε στο πλαίσιο των ειδικών οδηγιών για το χρηματοπιστωτικό τομέα, είτε στο πλαίσιο των μελλοντικών διατάξεων τη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και τέλο, αλλά είναι και εξίσου σημαντικό με τα προηγούμενα, ελπίζω τα επόμενα βήματα τη Κομισιόν να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών, το οποίο τελικά θα μπορούσε να οδηγήσει στην πλήρη εναρμόνιση των κανονισμών ε, περί προστασίας των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κυρία Πιατικάινεν. Περνάμε τώρα στις πολιτικές ομάδες.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 questo fondamentale intervento di armonizzazione è una condizione sine qua για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, την βελτίωση των, ε, της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Εδώ και ένα χρόνο ο καθηγητής κ. Μόντι έλεγε στην έκθεσή του προς, προς τον πρόεδρο Μπαρόσο ότι ο καταναλωτής και η ευημερία του καταναλωτή είναι ο στόχος της εσωτερικής αγοράς. Ο νομοθέτης λοιπόν θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία σχετικά με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και έτσι να δοθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στο λιανεμπόριο. Η ρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται πλήρως σε σχέση με τις προσδοκίες του κοινού και είμαι πεπισμένος ότι ο Επίτροπος ΣΒΑΜ θα επιδείξει τις ικανότητες που απαιτούνται τις διαπραγματευτικές και θα καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για δυόμιση λεπτά έχει το λόγο η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι ήταν σκληρές οι διαπραγματεύσεις που υποχρεωθήκαμε να διεξαγάγουμε γιατί υπήρχαν αποστάσεις ανάμεσα στις απόψεις μας κύριε Σφάπ στην αρχή της συζητήσεως και δεν ήταν διόλου απλό και εύκολο να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Ωστόσο, στις διαπραγματεύσεις αυτές επιτύχαμε να επιφέρουμε σημαντικές βελτιώσεις. Μάλιστα και μετά την ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που εν τέλει επιτρέπουν και στην δική μου πολιτική ομάδα να υπερψηφίσει το πακέτο αυτό συμβιβασμών. Και γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό μετά από τις συζητήσεις που διεξαγάγαμε. Όντως επιφέραμε βελτιώσεις. Η ελάχιστη εναρμόνιση λοιπόν τώρα αποτελεί και πάλι βάση της οδηγίας με εξαιρέσεις για περιστάσεις που δεν εναρμονίζονται. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, τυχερά παιχνίδια, τα αφήσαμε εκτός του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας, διότι πρόκειται για τομείς που απαιτούν ειδική ρύθμιση, ειδικού κανόνες. Δεν μπορούν να ενταχθούν ή να υπαχθούν στις συνήθεις ρυθμίσεις. Επίσης, υποχρέωση ενημέρωσης απέναντι στους πολίτες, απέναντι στους καταναλωτές. Αυτή η να υπαχθουν στις συνηθει ρυθμισεις επισης υποχρεωση ενισχύθηκε σημαντικά και γι' αυτό η διαγραφή του κεφαλαίου 2, αγαπητή Προεδρεύουσα, θα ήταν ακριβώς η διαγραφή αυτών των υποχρεώσεων. Αυτό δεν πρόκειται να υποστηρίξουν οι σοσιαλδημοκράτες ποτέ. Περιλάβαμε και τα ηλεκτρονικά προϊόντα στο πεδίο εφαρμογή που αρχικά δεν προβλέπονταν. Ειδικά όμως για το εμπόριο από μακριά με το διαδίκτυο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και στην τελική ευθεία επιτύχαμε να βελτιώσουμε πολύ και τις πωλήσει που γίνονται από πόρτα σε πόρτα. Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να υπερψηφίσουμε. Δεν κρύβω όμως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα και ιδίω σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 5, καταχρηστικές ρήτρε δηλαδή, όπου διόλου δεν μα ικανοποιεί και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και αν αυτό καταστεί απαραίτητο δεν θα το υποστηρίξουμε καθόλου. Επίσης οι υπηρεσίες οικονομικού χαρακτήρα έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση ενημέρωσης. Εδώ πιστεύω ότι σημειώνονται πολύ σημαντικά προβλήματα. Εδώ κυρία Επίτροπε θα χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε. Διότι στην δική σας αρχική πρόταση περιλαμβάνονταν και εγώ νομίζω ότι πρέπει να περιληφθούν. Εν συμπεράσματι θα υποστηρίξουμε την δέσμη των συμβιβαστικών προτάσεων θα ζητήσουμε να γίνει η εκ νέου παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε συμφωνήσει να ολοκληρωθεί η πορεία στην πρώτη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ για τους Μακράτες ε, και φιλέτερους. Ο κύριος Ροσφόρ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Αγαπητοί ε, Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, είναι σημαντικό το κείμενο, δεν αποτελεί επανάσταση, δεν θα πούμε ότι όλα ήταν χάλια πριν και όλα είναι τέλεια τώρα. Παρ' όλα αυτά, το κείμενο συνιστά σημαντική πρόοδο σε αυτό βέβαια το προσωρινό στάδιο των εργασιών μας. Το βασικό στοιχείο είναι η καλύτερη πλαισίωση των εξαποστάσεων ε, πωλήσεων και ιδίως στο διαδίκτυο. και Κεφάλαιο 3 Πρέπει να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα αυτό. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πολύ χρήσιμο, διότι διευρύνει την επιλογή του καταναλωτή, του επιτρέπει να βρει φθηνότερα τα προϊόντα και επιτρέπει επίση στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, στου βιοτέχνε να βρουν νέε διεξόδου, νέε αγορέ. Θα έπρεπε λοιπόν για να προοδεύσουμε στον τομέα αυτό να το κάνουμε με ευρωπαϊκό τρόπο, δηλαδή να είναι πάρα πολύ στοχευμένη η προσέγγιση μα και να προχωρήσουμε σε πλήρη εναρμόνιση και των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων όλων των πλευρών. Θα έπρεπε, παραδείγματο χάρη, ένα Ιταλό πελάτη που αγοράζει σε ένα βελγικό-γερμανικό site να ξέρει ότι από εδώ και πέρα θα έχει τα ίδια δικαιώματα, την ίδια προστασία. Αυτό θα καταστήσει δυνατό αυτή η οδηγία. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί μέσα σε 14 μέρες πλέον σε όλη την Ένωση να υπαναχωρήσει. Θα ξέρει δηλαδή ακριβώς το σύνολο που θα πρέπει να καταβάλει και δεν θα τον περιμένει εκ των υστέρων ε, κακή έκπληξη. Άρα με ένα διπλό κλικ θα μπορεί να επιβαληθεύσει την παραγγελία του σε κάθε περίπτωση. Σίγουρα κάποιες ε, συμπεριφορές ε, θα αλλάξουν άρδιν και κάποιες φορές σημαντικό ποιε θεωρούνται διατάξει κάποιων χωρών που δεν υπάρχουν καν σε άλλε χώρε. Θα πρέπει να αλλάξουν κάποιε συμπεριφορέ υπέρ του γενικότερου συμφέροντο των καταναλωτών. Πρέπει να είμαστε σαφεί. Επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση στο κείμενο και θα πρέπει να το κάνουμε και στο μέλλον μαζί με το Συμβούλιο και μαζί με την Κομισιόν. Χαίρομαι γιατί έγιναν κάποια ανοίγματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήδη έχουμε κάνει σημαντική δουλειά χάρη στον εισηγητή μας, τον Αντρέα Σβά, που θέλω θερμά να τον ευχαριστήσω. Όμως ο πραγματικό ε, καρπό αυτών των προσπαθειών είναι να υπερψηφιστούν αύριο τροπολογίε από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Διότι είναι πολύ εύθραυστη η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην νέα αγορά και χρειάζεται πολιτική βούληση για να την ε, διατηρήσουμε και ελπίζουμε να την ενισχύσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ροσφόρ. Από την ίσια ο κύριος Μπίλαν δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντα θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σφαμπ. Προσπάθησε πολύ και συνεργάστηκε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με πολύ καλό τρόπο με όλους τους ενδιαφερομένους. Ελπίζουμε ότι η τελική μορφή της συμφωνίας θα οδηγήσει σε ε, μια ασφάλεια τους καταναλωτές σχετικά με τις αγορές εξ και ιδιαίτερα τις αγορές μέσω διαδικτύου. Ελπίζω με τη νέα οδηγία ο καταναλωτής να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις αγορές εξ και ελπίζω οι κανόνες και οι εγγυήσει να ξεκαθαριστούν καλύτερα. Η εναρμόνιση ανάμεσα στις διάφορες χώρες για τέτοιου είδους συναλλαγές είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο και νομίζω ότι αυτό θα ενθαρρύνει και περισσότερες επιχειρήσεις να ενταχθούν σε τέτοιου είδους συστήματα πωλήσεων, ενισχύοντας έτσι την εσωτερική αγορά. Ελπίζω λοιπόν η κατάληξη των προσπαθειών να ενισχύσει τις πωλήσει online και να ωφελήσει τον ανταγωνισμό. Πρώτον, αυτό το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε είναι ένα κείμενο ισόρροπο, ένα κείμενο το οποίο να προστατεύει με τον ίδιο τρόπο τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην φύγει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, μέχρι τώρα έχουμε διαπραγματευτεί, θα έλεγα, στον τομέα της εναρμόνισης ένα κείμενο το οποίο θα χαρακτήριζα πραγματιστικό Έχουμε λοιπόν ήδη διασφαλίσει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και πρέπει να γίνει καλύτερο. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις ε, πωλήσει και τις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Έχει γίνει διαπραγμάτευση και σχετικά με το κεφάλαιο 5 και έχουν γίνει κάποιες προτάσεις, διατυπωθεί κάποιες προτάσεις σχετικά με την διαπραγμάτευση των συμφωνιών και των συναλλαγών και την αποφυγή καταχρήσεων από πλευρά των επιχειρηματιών. Είναι κρίμα που είναι σε, είναι εκκρεμότητα το τελικό κείμενο, δεν είναι έτσι κι αλλιώς ένα τέλειο κείμενο. Ελπίζω όμως ότι σε μια δεύτερη διαπραγματευτική φάση θα καταφέρουμε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο και για τους καταναλωτές και για τους επιχειρηματίες. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπίλαν. Εξ ονόματος των Πρασίνων, η κυρία Τουρούνεν για δύο λεπτά. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Στο σχέδιό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι οι πολίτες εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να βρεθούμε στο επίκεντρο των εργασιών για την ενιαία αγορά. Αυτό είναι σημαντικό. Όταν αύριο θα ψηφίσουμε την οδηγία επί της οποίας εργαζόμαστε ήδη από χρόνια. Το κείμενο που θα ψηφίσουμε αύριο, όπως γνωρίζουμε, έχει τροποποιηθεί σημαντικά. Ξεκινώντας από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μαρτίου 2008. Ρίξαμε το βάρος μας ιδίως στους τομείς εκείνους όπου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές αλλά και για την οικονομία. Οι χώρες μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν και αυστηρότερους κανόνες όπου αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Για παράδειγμα, τροποποίησης υπέρ των καταναλωτών όταν αγοράζουν μέσω διαδικτύου. Υπάρχουν κοινοί κανόνες, υπάρχουν ορισμένες καινοτομίες και δίνω ορισμένα παραδείγματα. Ως καταναλωτής μπορεί να έχει δικαίωμα ανακλήσεως εντός δύο εβδομάδων εάν αγοράσει κάτι από το διαδίκτυο. Επίσης η συνολική τιμή πρέπει να είναι σαφής για τον ε, καταναλωτή και τέλος πρέπει να είναι σαφή και τα στοιχεία του ε, εμπόρου. Δεν πρόκειται μόνο για εμπορεύματα τα οποία είναι ε, απτά, δηλαδή είναι πραγματικά αντικείμενα, αλλά πρόκειται και για άειλα αντικείμενα, όπω μουσική για παράδειγμα. Η πρόταση που θα κληθούμε να ψηφίσουμε αύριο δεν είναι τέλεια. Εμεί θα προτιμούσαμε μια ευρύτερη εφαρμογή οδηγία. Θα θέλαμε να δούμε να σημειώνονται πρόοδοι σε όλου του τομεί. Αλλά τέλο πάντων η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Και μάλλον στη στιγμή αυτή αυτό φαίνεται πω είναι το εφικτό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταρρύξει σε ένα καλό, λογικό αποτέλεσμα υπέρ των καταναλωτών. Ευχαριστώ εκ μέρου τη ε, ΓΚΟΕ, ΕΝΤΖΕΛ. Για 1,5 λεπτό έχει το λόγο ο κύριο Τριανταφυλλίδη. Κύριε Πρόεδρε, ω πολιτική ομάδα είχαμε θέσει από την αρχή την αποφυγή μείωση στα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχική πρόταση τη Κομισιόν, αν και ιδιαίτερα φιλόδοξη, αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύναμη για να καλύψει τι ανάγκε του συνόλου των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό η πρόταση για μια πλήρω εναρμονισμένη οδηγία ήταν κόκκινη γραμμή και έγινε σαφές ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με χαμηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην εε. δύο στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την πρόταση του κοινοβουλίου για την οδηγία. έχουμε μπροστά μας μια εντελώς νέα πρόταση από το κοινοβούλιο πολύ διαφορετική από αυτή που προτείνεται από την επιτροπή και με διαφορετική προοπτική από το συμβούλιο ο πυρήνας της πρότασης αυτής είναι η μεικτή προσέγγιση στο επίπεδο της εναρμόνισης αφήνοντας τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ορίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές όταν το αποφασίζουν. το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. επιμείναμε από την αρχή ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες οι υπηρεσίες υγείας και τα τυχερά παιχνίδια θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας καθώς δεν είναι σχετικές με τις σχέσεις έμπορος καταναλωτής και έχουν διαφορετική προσέγγιση. Είμαστε ικανοποιημένοι ότι αυτό λήφθηκε υπόψη. Με την υποστήριξη της πρότασης του Κοινοβουλίου δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ότι στηρίζουμε ανεφόρον την πρόταση της Κομισιόν. Αντίθετα, επιδιώκουμε μια ισχυρή συνεχτική θέση και καλούμε τη Κομισιόν αλλά και το Συμβούλιο να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τον πυρήνα της πρότασης του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τον βαθμό εναρμόνισης και τις λοιπές διατάξεις για τις συμβάσεις πώλησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τριανταφυλλίδη. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Ρώση για 1,5 λεπτό. Τα δικαιώματα των πελατών θα έλεγα όπως λέγεται στα αγγλικά customer rights είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και πρέπει να του δώσουμε ε, πολύ μεγάλη σημασία και σε πολιτικό επίπεδο και σε νομικό επίπεδο. Η τροπολογία μας για το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος σαν παράδειγμα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τελικά τον καταναλωτή χωρίς να θίξει τον επιχειρηματία. Το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να καταργήσει ε, και να ακυρώσει τα θετικά στοιχεία τα οποία οι πολιτικές ομάδες έχουν συνεισφέρει στην πρόταση της Επιτροπής. Αν επιμείνει το Συμβούλιο προς την κατεύθυνση αυτή θα καταψηφίσουμε την πρόταση. Και η ευθύνη δεν θα είναι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Υπάρχουν θέματα εναρμόνισης, υψηλότερης εναρμόνισης, όπου η Λέγκα Νόρντο θα συμφωνήσει. Αλλά αυτό μόνο αν βοηθάει τον καταναλωτή και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένα περίπλοκο θέμα το θέμα της προστασίας του καταναλωτή και γι' αυτό από την αρχή έπρεπε να έχουμε λάβει υπόψη όλους τους καθοριστικούς παράγοντες που δεν το κάναμε. Δεν πρέπει να επανερχόμεθα σε θέματα τα οποία έχουν επιληθεί και ξεπεραστεί και νομίζω ότι θα πρέπει να δεχθεί τις τροπολογίες από τις πολιτικές ομάδες ως έχουν το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των ο κύριος Όμπερ Μάγερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολο, για παράδειγμα, για τον καταναλωτή το κατέβασμα άϊλων ε, περιεχομένων από το διαδίκτυο για παράδειγμα με συνδρομές. Εδώ χρειάζεται λοιπόν ασφαλώς ένα νομικά προβλεπόμενο δικαίωμα ανάκλησης. Το ίδιο για τις πωλήσει από πόρτα σε πόρτα, όπου συχνά ε, υφίστανται σημαντικές πιέσεις οι καταναλωτές. Άλλη περίπτωση είναι όταν προσκαλείται από τον καταναλωτή στο σπίτι του κάποιος για να επισκευάσει κάτι. Χρειαζόμαστε λοιπόν ρυθμίσεις, πραγματική προστασία των καταναλωτών, αλλά ταυτόχρονα προστασία των συμφερόντων των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Σας ευχαριστούμε κύριο Μπερμάγερ. Περνάμε στους λοιπούς ομιλητές. Για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Κοράτσα. Η συμβιβαστική πρόταση που έχουμε μπροστά μας είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός. Ελπίζω να καταλήξουμε και στο θέμα του δικαιώματος επιστροφής και επίσης στο θέμα της παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όμως το Συμβούλιο να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα για να αντιμετωπιστούν τα θέματα των καταχρηστικών ρητρών και νομίζω ότι ασχολούμαι με το θέμα εδώ και αρκετά χρόνια και ζητώ να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση. Είμαι πεπισμένη ότι οι κοινοί κανόνες είναι θετικοί και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές και για τον ανταγωνισμό, την νομική βεβαιότητα, την ασφάλεια του καταναλωτή και τη μείωση των τιμών. Πρέπει λοιπόν να ισορροπήσουμε το κείμενο ανάμεσα στο χαμηλό κόστος για τις επιχειρήσεις και το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Δεν θα πρέπει εμείς να συνεχίζουμε μια λογική αντιπαράθεση ανάμεσα στους καταναλωτές και τους πολιτές. Νομίζω ότι οι κοινοί κανόνες θα βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτές τις λανθασμένες εικόνες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει ε, να μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στους καταναλωτές. Μέχρι τώρα δυστυχώς το Συμβούλιο έχει περιορίσει τη συζήτηση σε μια προσπάθεια ουσιαστικά συγκριτικού δικαίου και σε μια στήρα αντιπαράθεση η οποία δεν υπηρετεί το κοινό συμφέρον των Ευρωπαίων. Αυτό θα πρέπει να κυριαρχήσει. Νομίζω ότι οι εθνικές εξαιρέσεις όπως τις επιζητούν οι σοσιαλδημοκράτες εμποδίζουν τους πολίτες να εκμεταλλευτούν πλήρως την κοινή αγορά σε μια περίοδο κρίσης με αυξανόμενο τον προστατευτισμό είναι εύκολο αλλά και ανεύθυνο το να είναι κανείς λαϊκιστής. Υποστηρίζω τον ΣΦΑΜ για μια εξαιρετική δουλειά και τον συγχαίρω για μια ακόμη φορά και ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσει θα πάνε καλά. Νομίζω ότι η οδηγία για τους καταναλωτές θα είναι καταληκτικό σημείο της προσπάθειας ανάκαμψης της αγοράς, ενίσχυσης της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Σας ευχαριστούμε κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Μασίπ. Υπάρχουν σημαντικά σημεία τα οποία επιδέχονται βελτίωση. Γι' αυτό και πρέπει να αναπέμψουμε την έκθεση στην Κομισιόν. Η πρόταση αρχική ήταν κακή. Μας το έλεγαν οι ενώσεις καταναλωτών σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. και ειδικά οι Ένωση Καταναλωτών ε, του Αστούρια και του Προέδρου της του του μου το είχαν πει. Η Γενική Αρχή μιας μέγιστης εναρμόνισης ε, του άρθρου 4 ε, ήταν κάτι που δεν έπρεπε να το δεχθούμε. Πρέπει να πω ότι η μέγιστη εναρμόνιση για να έχουμε την ίδια προστασία σε όλα τα κράτη-μέλη προϋποθέτει και συνεπάγεται την μείωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Υπάρχουν όμως μεγαλύτερες παραδόσεις προστασίας ε, των καταναλωτών σε κάποιες χώρες. Και γι' αυτό θέλω να τονίσω σε κάθε περίπτωση ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και οι συμβατικέ καταχρηστικέ ρήτρε ε, να μην περιληφθούν σε έναν κατάλογο εξαντλητικό ώστε να μπορεί κάθε κράτο μέλο να αυξήσει τι ρήτρε, τον αριθμό των ε, ρητρών ή ε, να ακυρώσει αυτέ που θεωρεί απαράδεκτε για την προστασία των καταναλωτών. Και θα πρέπει να δοκιμάσουμε τι μεμονωμένε ρήτρε, να τι ελέγξουμε. Γιατί οι έμποροι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι έγινε ιδιωτική διαπραγμάτευση μία ε, των ρητρών. Οι συμβατικέ ρήτες πρέπει να εκφράζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο και είμαστε κατά του να υπάρχει, επαναλαμβάνω, μέγιστη εναρμόνιση σε σχέση με τι καταχρηστικέ ρήτρε. Το Ευρωβαρόμετρο μα λέει ότι το 79% των εμπόρων πιστεύουν ότι η πλήρη εναρμόνιση στον τομέα αυτό δεν θα έχει πολύ λίγο ή καθόλου αποτέλεσμα. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για δυόμιση λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Χάρμπορ. Κανονικά θα έπρεπε να είχα περισσότερο χρόνο γιατί πολλοί συνάδελφοι δεν είναι παρόντες. Σε πάση περιπτώσει θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη τα οποία προσπάθησαν προς την κατεύθυνση αυτή με την καθοδήγηση του ΣΒΑΜΠ. Ήταν μια ισχυρή ομάδα με τους σκιώδεις εισηγητές και προσπαθήσαμε με πολύ ενδιαφέρον και εμπειρογνωμοσύνη να κάνουμε βήματα πρόοδου σε ένα δύσκολο τομέα. Όπως είπε η Βιβιάν Ρέντινγκ, τώρα πλέον θα πρέπει οι συνομοθέτες να προχωρήσουν και να καταλήξουν σε αποφάσεις. Ο χρόνος που χρειάστηκε για να φτάσουμε εδώ υποδεικνύει, αν θέλετε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε πολιτικά και σε επίπεδο Συμβουλίου και σε επίπεδο Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο όμως, όπως και σε άλλα θέματα στο παρελθόν, επέδειξε ότι έχει την ικανότητα να λειτουργήσει με πνεύμα συμβιβαστικό. Γι' αυτό λοιπόν αύριο σωστό θα είναι να ψηφίσει το Κοινοβούλιο τις τροπολογίες, να στείλει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα σχετικά με το τι επιθυμούμε και να, παραπέμψουμε, και να μην παραπέμψουμε το θέμα εκ νέου στην Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Προεδρία η οποία είναι δεκτική και θα εξετάσει τις θέσεις μας μετά από τις αλλαγές οι οποίες θα υπάρξουν. Θα θέλαμε να κλείσουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις, αλλά από την άλλη θέλουμε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να βρουν μια πλατφόρμα στο εσωτερικό της οποίας να μπορέσουν να συζητήσουν για να λύσουν τις διαφορές. Πρώτον, εγώ θαυμάζω τον ενθουσιασμό της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι η οδηγία αυτή είναι πράγματι τόσο σημαντική. Είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο αν θέλετε, ένα πέρασμα. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα πρώτο προσεκτικό βήμα για την εναρμόνιση ενός θέματος που προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα και πολλή πολιτική αναταραχή είναι κατανοητό οι καταναλωτές και οι οργανώσεις τους να μην θέλουν να τους αφαιρούνται δικαιώματα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι η συμβιβαστική πρόταση προσθέτει αξία και για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο και το εμπόριο ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες. Τέλος, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πω το εξής. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για περισσότερη εναρμόνιση. Έχουμε πάρα πολλές πολυδιασπασμένες πρωτοβουλίες και οι δική σας και για τις ε, ε, συμβάσεις και απαιτείται ένα, μια προσπάθεια στρατηγική μακροπρόθεσμη έτσι ώστε να συμπληρώσουμε τα ενδιάμεσα βήματα. Ευχαριστώ κύριε Χάρμπορ. Για δύο λεπτά. Η κυρία Χάνσλικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου Ανδρέας Σβάμπ για την σύνταξη της έκθεσης που δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τονίσαμε συχνά πόσο σημαντική είναι η οδηγία αυτή για τους καταναλωτές αλλά και για το εμπόριο, ιδίως το ηλεκτρονικό και τις διαμεθοριακές συναλλαγές οι καταναλωτές όταν αγοράζουν κάτι τι επιγραμμικά θέλουν εγγύσεις ότι πρώτον τα πράγματα που αγοράζουν, οι υπηρεσίες που αγοράζουν πραγματικά θα παρασχεθούν. Αναμένουν ποιότητα. Γι' αυτό και πρέπει να εξασφαλίσουμε βεβαιότητα και ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Αλλά και οι επιχειρήσεις αναμένουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο δεν θα είναι επιβαρυντικό για αυτές. Κατά τη γνώμη μου έχουμε πλησιάσει τώρα τον στόχο αλλά δεν τον έχουμε ακόμη επιτύχει. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα επωφεληθούν περισσότερο από μια συνολική εναρμόνιση Ιδίω στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πάντως σε πολλού τομεί κλειδιά βρήκαμε λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες των καταναλωτών και συμφιλιώνουν τις ανάγκες αυτές ή τις λύσεις που δίνονται και με τα ενδιαφέροντα των επιχειρηματιών. Από την άλλη μεριά βρίσκω σωστή και την τροπολογία που δίνει στον έμπορο την δυνατότητα να, που προσφέρει μάλλον στον ε, καταναλωτή τη δυνατότητα να ζητήσει αποδείξεις. Νομίζω ότι είναι μια σωστή προσπάθεια και μια σωστή προσέγγιση. Σα ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό έχει το λόγο κυρία Βερνιό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Σφαπ καθώς και όλους τους σκιώδεις εισηγητές, ιδίως την Εύελιν Κέπχαρτ για το έργο που έχουν επιτελέσει. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν πράγματι ήταν παράλογη και έθετε σε κίνδυνο το επίπεδο της προστασίας των καταναλωτών θέλοντας να προβεί σε μια πλήρη εναρμόνιση. Αυτό όμως ε, μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο αν η εναρμόνιση γίνει προς τα πάνω και προς τα κάτω, όπως πρότεινε η Κομισιόν. Χαίρομαι λοιπόν για τις περισσότερες από τις συμβαστικές προτάσεις, οι οποίες ε, σέβονται τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να μπορούν να εισαγάγουν, αν το επιθυμούν, πιο αυστηρούς κανόνες, εγγυόμενα ένα κατώτατο, υψηλό όμως επίπεδο ε, για ε, όλους τους καταναλωτές της Ένωσης. Επομένως, η σύμβαση μέγιστη μπορεί να διαρκέσει 12 μήνες, βελτιώνονται οι όροι για τις εξαποστάσεως ε, ή εκτός καταστήματος πωλήσει και υπάρχει και αυτή η προθεσμία για την ανάκληση ε, που γίνεται 14 ημέρες. Αλλά η εναρμόνιση η πλήρης ε, στο κεφάλαιο 5 είναι απαράδεκτη. Μιλάω για τις καταχρηστικές ρήτρε. Όχι μόνο το επίπεδο της προστασίας είναι ανεπαρκές, όπως προτείνεται εκεί, αλλά ουσιαστικά γνωρεί την πραγματικότητα των ε, ε, απατηλών δόλιων πρακτικών που υπάρχουν. Δεν μπορεί να ε, το επιτρέψουμε αυτό και είναι ανεύθυνο να εμποδίσουμε τα κράτη-μέλη να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν οι συνομοθέτες να καταλήξουν σε ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο θα εξασφαλίζει ένα κατώτατο κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών αλλά υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Σας ευχαριστούμε κυρία Βερνιό. Το λόγο για ένα λεπτό. Ο κύριο Κόζουσνικ. <clears throat> <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω το θαυμασμό μου για την δουλειά του κυρίου Σφαμπ, ο οποίος χρειάστηκε να αντιμετωπίσει 1.600 τροπολογίες και να μας παρουσιάσει μια πολύ ισόρροπη έκθεση έχει βελτιώσει τις βασικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλύτερη νομοθεσία, απλούστευση της νομοθεσίας, περισσότερες εγγυήσεις, λιγότερα εμπόδια στην εσωτερική αγορά για τους επιχειρηματίες. Και δεύτερον, σέβεται και την αρχή της μέγιστης δυνατής εναρμόνισης στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, με ελάχιστες εξαιρέσεις από πλευράς των κρατών μελών δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ακόμα σε πλήρη εναρμόνιση αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να αποσύρουμε τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ κύριε Κόσουσνικ. Λέχνα. Ευχαριστώ. Εγώ θα τονίσω ότι παρόλες τις πολλές βελτιώσεις που επιφέρθηκαν στην πρόταση της Κομισιόν και που αυτά το οφείλουμε κυρίως στον Ανδρέα Σφάπ θεωρώ ότι το πακέτο που βάλετε εν τέλει έχει τόσες υπερβολικές ρυθμίσεις που θα, είναι, θα επιβαρύνουν σοβαρά το έργο των μικρών και μισών επιχειρήσεων χωρίς να προστατεύουν πραγματικά τον καταναλωτή. Και δεν προωθούν την υπόθεση της νέας αγοράς. Λόγω του πολύ σύντομου χρόνου που διαθέτω θα αναφερθώ μονάχα σε ένα θέμα. Η πρόταση της Κομισιόν διεύρυνε συνολικά δύο ορισμούς. Φάνηκε άλλωστε και με τις 1600 αυτές τροπολογίες ότι ήταν αδύνατο να γίνει μια λογική συζήτηση στο Κοινοβουλίο. Για αυτές τις διευρύνσεις των ορισμών δεν προσφέρθηκε άλλωστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καμία αιτιολόγηση. Αφενός η συνθήκη για, η, συγγνώμη, η σύμβαση πωλήσεων εξ αποστάσεως, εδώ επιφέρθηκαν κάποιες διορθώσεις και τις καλωσορίζω. Το δεύτερο όμως είναι, και αυτό με απασχολεί ιδιαίτερα, το εμπόριο εκτός χώρων επιχειρήσεων. Στο μέλλον κάθε σχετική σύμβαση θα επιβαρύνεται με διατάξεις, με δικαιώματα ανακλήσεως, ακόμα και αν ο καταναλωτής έχει ζητήσει να έρθει στο σπίτι του ο ελαιοχρωματιστής ή ο μαραγκός. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, πάλι χάρη στον Αντρία Σουάμπ εδώ έγιναν πολλές βελτιώσεις, παρόλα αυτά παραμένουν τόσες πολλές παγίδες που θα είναι μοιραίες για μικρές επιχειρήσεις. Αυτό το τμήμα της προτάσεως κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως περιττό και θα μπορούσε μια χαρά να διαγραφεί. Επίσης τα κεφάλαια 4 και 5 θα μπορούσαν να διαγραφούν. Τα υπόλοιπα νομίζω είναι ανεκτά. Ευχαριστώ κύριε Λέχνερ. 1,5 λεπτό. Η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή κύριο Σουάμπ και τη σκιώδη σοσιαλίστρια εισηγήτρια κυρία Γκέπχαρτ να τους ευχαριστήσω και ταυτοχρόνως να τους θαυμάσω γιατί είχαν πάρα πολύ επιμονή αλλά και εξαιρετικά μεγάλη υπομονή για να μας οδηγήσουν σε αυτό το σημείο το οποίο συζητούμε σήμερα και το οποίο δίνει νομίζω μια καλή βάση εργασίας και στην επίτροπο ρέντινγκ που εκφράστηκε κατά τη γνώμη μου με έναν τρόπο που μας επιτρέπει να έχουμε αισιοδοξία προσωπικά θεωρώ την ελάχιστη εναρμόνιση μια πολύ καλή και ταυτοχρόνως ρεαλιστική βάση για να εργαστούμε. προέρχομαι από ένα κράτος την ελλάδα που έχει επιτύχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο διασφάλισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών και όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα ήθελα αυτό το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών να πηγαίνει προς τα κάτω ομολογώ ότι προβληματίστηκα εξαιρετικά όταν άκουγα για πρώτη φορά και τα επιχειρήματα του κυρίου σουαμπ για την μέγιστη εναρμόνιση. εκεί όμως πραγματικά ήρθε στο μυαλό μου κάτι που είχα διαβάσει σε ένα περιοδικό. κάποιος προσπάθησε να φτιάξει το ωραιότερο γυναικείο πρόσωπο παίρνοντας τα μάτια μιας ηθοποιού τη μύτη μιας τραγουδίστριας τα χείλη μιας άλλης ηθοποιού στο τέλος το πρόσωπο που βγήκε ήταν ένα τερατούργημα. κάνω αυτήν την ε, παρομοίωση για να δείξω ακριβώς ότι μπορεί να ξεκινάμε με τις καλύτερες των προθέσεων αλλά να μην καταλήγουμε στο ποθητό καλό αποτέλεσμα. γι' αυτό λοιπόν κλείνω κύριε πρόεδρε θεωρώ ότι η ελάχιστη εναρμόνιση είναι η σωστή βάση εργασίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Αράπτη. Για δύο λεπτά ο κύριος Άμπατ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντρέα Σουάμπ. Μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε μια ευρύτατη συμφωνία ανάμεσα σε πολιτικές ομάδες που δεν το προβλέπαμε στην αρχή. Η Ευρώπη πρέπει να είναι συγκεκριμένη, πρέπει να είναι προοδευτική και θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν μια σύμβαση αγοράς όταν δουν ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους η αγορά τους. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τις συμφωνίες πλαίσιο, πρέπει να ενισχύσουμε τις αγορές ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες αγοράς στις διάφορες χώρες. Θα πρέπει να εξορθολογήσουμε την εσωτερική αγορά. Ξέρετε ότι μόνο το 22% των αγορών στην Ευρώπη είναι διασυνοριακές, είναι από διαφορετικές χώρες και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πρέπει να φανούμε φιλόδοξοι, πρέπει να φανούμε πραγματιστές, να μην υπάρχει εναρμόνιση αν δεν υπάρχει αντίστοιχη προστασία. Γι' αυτό ακριβώς χαίρομαι που μπορέσαμε να συγκρατήσουμε κάποια τμήματα των εθνικών νομοθεσιών στα οποία εμένουν οι χώρες. Για τη Γαλλία οι καταναλωτές μας θα συνεχίσουν να έχουν τις εγγυήσει για κρυφία ελαττώματα και ταυτόχρονα θα ρυθμιστεί το θέμα των πωλήσεων κατοίκων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δεξιά και η αριστερά πτέρυγα θα αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών. Ναι μεν περισσότερη Ευρώπη αλλά όχι η αδίποτε Ευρώπη. Μια Ευρώπη που να προστατεύει, να ε, διασφαλίζει, να παρέχει εγγυήσεις στους καταναλωτές, στους αγοραστές και στις επιχειρήσεις. 1,5 λεπτό η κυρία Σεχνάλοβα. Είχε ξεκινήσει η συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παλιά λέγαμε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα παρότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες να προστατεύουμε τους καταναλωτές, τους πελάτες. Ε, η ικανοποίηση του πελάτη δεν φαίνεται όμως να είναι ο στόχος, ο βασικός των επιχειρήσεων. Και γι' αυτό ακριβώς οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις έχουν μεγάλη σημασία και δεν θα πρέπει να μειώσει τα επίπεδα της προστασίας του καταναλωτή. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις διάφορες χώρες είναι διαφορετική. Πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στις χώρες όπου δεν υπάρχει ή υπάρχει σε χαμηλό επίπεδο νομική βεβαιότητα και υπάρχουν απειλές και εμπόδια για την εσωτερική αγορά. Εκεί όμως όπου η προστασία του καταναλωτή είναι αναπτυγμένη πρέπει να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για την τεράστια δουλειά που έκαναν. Η προστασία του καταναλωτή δεν είναι εις βάρος των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Κυρία Μπάστος, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε, συνάδελφοι. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Σφάμπ. Έχει διαπραγματευτεί τη συμβιβαστική πρόταση με πολύ σκληρό και ικανό τρόπο. Εμείς δεν θέλουμε μόνο να παρέχουμε υψηλά επίπεδα προστασίας στους καταναλωτές στην Ευρώπη, αλλά θέλουμε ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες και αγαθά σε όλες τις χώρες χωρίς μη απαραίτητες νομοθετικές παρεμποδιστικές ρυθμίσεις. Κάποιες νομικές ρυθμίσεις σήμερα κάνουν πολύ δύσκολο το διαμεθοριακό εμπόριο και αυτό δημιουργεί προβλήματα συνολικά στην εσωτερική αγορά Πρέπει λοιπόν το εμπόριο να γίνεται με σωστές συνθήκες, να είναι κατανοητή η σύμβαση αγοράς και θα πρέπει να εγγυηθεί την ποιότητα του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας ο έμπορος. Σχετικά με τις ε, αγορές μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου, τα προϊόντα και οι οδηγίες που παρέχονται θα πρέπει να είναι κατανοητές στους ε, καταναλωτές. Ελπίζω εν πάση περιπτώσει να καταλήξουμε σε μια ρύθμιση για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική οικονομικά. Ο κύριο Σάντσε Περισσέδο για δύο λεπτά. Αγαπητέ Πρόεδρε, το να έχουμε μια οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών το να έχουμε ένα οριζόντιο εργαλείο που θα πλουστεύει και θα συμπληρώνει τις τέσσερις οδηγίες είναι θετικό. Μια εσωτερική αγορά που θα χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή είναι σημείο κλειδί για την ανάπτυξη και τη βιώσιμη ε, απασχόληση. Δεν θα πρέπει βέβαια να παρεμποδίζεται η υιοθέτηση από τα κράτη-μέλη μέτρων τα οποία αυξάνουν την προστασία των καταναλωτών γιατί πλήρη εναρμόνιση πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις ε, που είναι απαραίτητο για να υπάρξει ένα συνεπές πλαίσιο σε διασυνοριακές ε, ε, συναλλαγές για να αποτελέσει προσθέμενη αξία. Το προβλέπει και η συνθήκη. Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων συμφωνούμε ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της πρότασης για να είναι πραγματικά οριζόντια και θα πρέπει να δούμε την ε, τομεακή και την κοινοτική αλλά ε, και την εθνική νομοθεσία ε, πώς θα απαλείψουμε κάποια κριτήρια εξειδίκευσης ή κάποια κενά. Δεν μας ικανοποιεί λοιπόν στο σημείο αυτό το κείμενο και θα πρέπει να έχει τελειοποιηθεί προτού γίνει η τελική νομοθετική πρόταση και θα πρέπει να έχουμε και έναν ευρωπαϊκό χάρτη των καταναλωτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ κύριε Σάντσεφ Πρεσέδο. Ο κύριος Μέσαρος, για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο ΣΒΑΠ για την δουλειά που έκανε. Η εναρμόνιση των κανόνων θα πρέπει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά και να φέρει ασφάλεια δικαίου. Αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις εκείνες, τις εταιρείες εκείνες οι οποίες θέλουν να προβούν σε διαμεθοριακές συναλλαγές. Η πρόταση του κ. Σφάπ να υπάρξει μια ελάχιστη εναρμόνιση δηλαδή και μια πλήρη εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών είναι και η μόνη αποδεκτή λύση. Ένα συνδυασμό ελάχιστη και πλήρου εναρμόνισης μπορούν να ικανοποιήσουν ω λύσει όλου παρεμποδίζονται οι διαμεθοριακές συναλλαγές αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο δεν επιτρέπει και την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. Οι στατιστικές δείχνουν ότι πολλοί φοβούνται, είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις ε, αγορές μέσω του διαδικτύου. Οι κεντρικές και ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες χρειάζονται ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο διότι δεν έχουμε επαρκή ενημέρωση των καταναλωτών όπως υπάρχει σε χώρες, στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν πρέπει να κάνουμε τη ζωή των ΜΜΕ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πιο δύσκολη και να προωθήσουμε το εμπόριο στην ενιαία αγορά. Ασφαλώς και πρόκειται για προτεραιότητα και ιδίω τη Ουγγρικής Προεδρίας. Είναι μάλιστα και συμβολικό ότι λίγες ημέρες μόνο μετά την Παγκόσμια ημέρα των καταναλωτών ε, ψηφίζουμε αυτή την πρόταση για να εξυπηρετήσουμε εκατομμύρια καταναλωτών και επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ. Περάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Κέλλη, το λόγο για ένα λεπτό. Θέλω. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Σφάμπ για το πολύ σημαντικό έργο που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια. Θέλω να συγχαρώ και την Ουγγρική Προεδρία, γιατί και αυτοί κάνουν πολύ σημαντική δουλειά. Πρέπει να πω επίσης ότι και η Επίτροπος πάντοτε είναι παρούσα. Σίγουρα η εναρμόνιση είναι σημαντική, αλλά το θέμα είναι να σημειώσουμε πρόοδο. Έχουμε το δικαίωμα της ανάκλησης, της παναχώρησης και έχουμε και τις ρήτρε ευελιξίας, που δεν είναι ευελιξία στις εθνικές κυβερνήσεις. Αν κάναμε το ίδιο και σε άλλες οδηγίες, τότε θα το είχαμε καταφέρει και καλύτερα. Και επίσης Έχουμε τις οδηγίες ε, για τις υπηρεσίες για την προστασία των δεδομένων. Καλό θα ήταν ε, να γίνει μια ε, συνεργασία για να ομοιογενοποιηθούν κάπως αυτές οι τρεις εκθέσεις. Θα συνεργαστώ με τον κύριο Σφάπ. Κυρία Ιγκούγιν, έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Επιτρέψατε μου καταρχάς ε, να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Σβάπτη και την κυρία Γκέπχαρτ για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. Δεν μιλάμε για μεγαλύτερο προστατευτισμό. Αυτό που θέλουμε είναι να μην περισταλούν τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα των καταναλωτών σε ορισμένα Γιατί εάν θέλουμε να επιμείνουμε να έχουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά για τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, πρέπει παράλληλα να θεσπίσουμε μια εξισορρόπηση του υψηλού επίπεδου προστασίας των καταναλωτών αλλά και της πρόσπισης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αυτή η ισορροπία, αυτή η συμφιλίωση περνά μέσα από την κατώτατη, ελάχιστη εναρμόνιση και από τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να μπορούν να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν πρόσθετες ρυθμίσεις που θα βελτιώνουν την προστασία των καταναλωτών. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ε, να υπάρχει η έννοια αυτού του κοινού προτύπου που θα σημαίνει ότι πολλοί καταναλωτές και πολλοί χρήστες θα περιοριστούν ε, τα δικαιώματά τους. Μπορεί να έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, αλλά θέλω να επιμείνω ότι δεν θα πρέπει να περικοπούν τα δικαιώματα που έχουν ήδη ε, καθιερωθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος ε, Μπουσόη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον κύριο Σφάμπ και τους συνεισηγητές του και τους σκιώδεις εισηγητές για μια εξαιρετική δουλειά. Ήταν δύσκολο να εξισορροπήσουμε τα συμφέροντα και των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Η συμβιβαστική πρόταση είναι καλή και έχει μεγάλη σημασία για όλους τους καταναλωτές. Υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις όπως η σωστή ενημέρωση, όπως και το δικαίωμα ανάκλησης. Στο 22α υποχρεούται ε, να παρέχει υπηρεσίες ε, ο επιχειρηματίας που δεν προεβλέπονται στο παρελθόν. Μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα και με τα ψηφιακά λιγόμενα αγαθά ή προϊόντα Πάντως είναι θετικά, θετική συνολικά η πρόταση και ελπίζω να γίνουν οι τελευταίες απαιτούμενες ρυθμίσεις για να καταλήξουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριε Μπουσόη. Κυρία Τικάου, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε όλοι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της σωστής ενημέρωσης όταν υπογράφουν μια σύμβαση. Οι έμποροι θα πρέπει να ενημερώνουν σωστά τους καταναλωτές πριν συμφωνήσουν, ακόμα και για τις συνθήκες ε, κάτω από τις οποίες θα κρατηθούν χρήματα από την πιστοτική κάρτα του καταναλωτή. Πρέπει επίσης να προστατευτεί ο καταναλωτής από τις καταχρηστικές ρήτρες, Πολλές φορές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε πιστοτικές υπηρεσίες και σε ε, τέτοιου είδους υπηρεσίες δυστυχώς οι ρήτρε ε, είναι με πάρα πολύ μικρούς χαρακτήρες και αναγκάζονται οι πελάτες να υπογράφουν μια σύμβαση χωρίς να είναι σωστά ενημερωμένοι. Ακόμα και αν διαβάσουν τις ρήτρε αυτές και διαφωνούν δεν έχουν ουσιαστικά κανένα διαπραγματευτικό δικαίωμα. Η πρώτη επίπτωση είναι ότι το συμβόλαιο είναι ένα συμβόλαιο τύπος το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, έτσι λένε οι επιχειρήσεις. Ενώ ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να κάνει τις απαιτούμενες αλλαγές προστατεύοντας τα συμφέροντα του. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Για ένα λεπτό κυρία Ρόιτοβα. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Σφάπ για την θαυμάσια εργασία του και για την υποστήριξη που προσέφερε στις τροπολογίες μου που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να λαμβάνουν τα αγαθά που παραγγέλουν σε οποιαδήποτε χώρα μέλος. Ένα τρίτο των εμπόρων αρνούνται να αποστέλουν εμπορεύματα πέραν των συνόρων και κυρίως σε νέες χώρες μέλη. Θα εξασφαλιστεί τώρα με τον τρόπο αυτό η διαλειτουργικότητα με απλούς όρους συμβάσεων και επίσης η δυνατότητα των χωρών μελών να επεκτείνουν την προστασία και σε μη κρατικές οργανώσεις και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους σαφώς καθορισμένα δικαιώματα και αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί στην ενιαία αγορά. ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως προβλέπει η στρατηγική την Ευρώπη 2020, ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών εγγυάται και ποιοτικά προϊόντα, αλλά και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, για να είναι πιο αποτελεσματική η εσωτερική αγορά. Δεδομένων των ελάχιστων κανόνων που ισχύουν, όλα τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ε, τις εσωτερικές τους αρχές. Και νομίζω ότι αυτή ακριβώς ε, είναι η στάση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θέλουμε να υπάρχει αναρμόνιση και υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών, βελτιώνοντας ε, το επίπεδο προστασίας με την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών πρέπει να υπάρχει και ε, ένα σωστό σύστημα ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωση. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην κοινή αγορά και να υπάρχει ένα μεγαλύτερο κύκλο προϊόντων. Αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ την κυρία Ντάντσιλα. Τώρα για ένα λεπτό έχει το λόγο η κυρία Κάλπεξ. a jelenleg hatályos európai fogyasztói szabályok minimális harmonizációs Ευχαριστώ. Με βάση την τρέχουσα νομοθεσία υπάρχει μια κατώτατη εναρμόνιση. Τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν τους δικούς τους κανόνες, αλλά αυτό θέτει σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να χαιρετήσω την πρόταση του κυρίου ΣΒΑΠ. Μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων πλέον ήρθε η ώρα να φτάσουμε σε μια λύση. Όπως είπε και η κυρία Γκιόρη, η Ουγγρική Προεδρία σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί. Χρειαζόμαστε ένα υψηλό επίπεδο προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Πρέπει να είναι ενήμεροι οι καταναλωτές ώστε να μπορούν να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή και δεν θα πρέπει να φορτώνουμε με περισσότερη γραφειοκρατία τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Για να έχουμε ενιαία αγορά θέλουμε και ενιαία δέσμη μέτρων. Γι' αυτό πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Σα ευχαριστώ κυρία Γκάλ Πελτ, η κυρία Ρέντινγκ, Επίτροπο έχει το λόγο. Uh, Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερως επικοδομητική. Όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι απαιτείται να υπάρξει μια πιο επικοδομητική και πιο αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή και οδηγία για προστασία του καταναλωτή από ό,τι σήμερα συμφωνούν ότι δεν είναι τέλεια η προτινόμενη ρύθμιση, αλλά σίγουρα είναι καλύτερη από αυτήν η οποία βρίσκεται ισχύ η οποία έχει πάρα πολλά κενά και όλοι συμφωνούν σε αυτό. Ε, σπάνια έχω δει λοιπόν μια τέτοια ομοφωνία σχετικά με, την, με τα καλά λόγια που άκουσε ο εισηγητής και οι συνεισηγητές του. Ελπίζω η ομοφωνία αυτή να συνεχιστεί στο μέλλον. Τώρα ξεκινάμε μια προσπάθεια την οποία θα χαρακτήριζα πρωτότυπη αλλά και ταυτόχρονα μια προσπάθεια η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι θα πετύχουμε καλύτερες νομοθετικές ρυθμίσεις από ό,τι στο παρελθόν. Συνεπώς σας ενθαρρύνω όλους να βοηθήσετε τους εισηγητές σας και να ξεκινήσουν με ξεκάθαρη εντολή τις διαπραγματεύσεις. Ξέρω ότι η Ουγγρική Προεδρία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της έτσι ώστε αυτές οι προσπάθειες, οι πρωτότυπες, να στεφθούν από επιτυχία. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Αγγέρη, από την Ουγγρική Προεδρία έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί βουλευτές, θέλω και εγώ να συμφωνήσω με όσους είπαν ότι πρόκειται για μια εξαιρετική επικοδομητική συζήτηση. Η Ουγγρική Προεδρία θέλει να σας ευχαριστήσει για τη στήριξή σας και οι υπερογνώμονες θέλουν να σας ευχαριστήσουν και θέλω να σας πω ότι θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το ίδιο πνεύμα. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τους δίκαιους συμβατικούς όρους ε, ή τον κατάλογο των ε, καταχρηστικών ρητρών που είπατε να μην είναι εξο, εξαντλητικός, να μην είναι διεξοδικός. Θα έχουμε σύντομα ένα κατάλογο, ο οποίος είναι ενδεικτικός. Άρα θα υπάρχει προσθέμενη αξία σε μια νέα δέσμη καταλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αθέμητες πρακτικές και τους αθέμητους όρους συμβάσεων. Απλά δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση επειδή το Συμβούλιο ήταν αντίθετο. Η κυρία Γκάλ Πέλτς από τη χώρα μου είπε για τη σημασία που έχει να καταλήξουμε σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να σας πω ότι επί Γαλλικής Προεδρίας δύο χρόνια πριν ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Είχαμε πάνω από 60 ομάδες εργασίας για το θέμα αυτό και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο ελιγμών πλέον για να, να μην υπάρχει αυτή η μειοψηφία εμπλοκή και εξού και αποφασίσαμε να περιορίσουμε το εύρο της οδηγίας, κυρίω εξ εξαποστάσεω ε, και εκτό καταστήματος πωλήσει. Παρά τώρα αυτό το περιορισμένο, ε, μάλλον με το περιορισμένο αυτό πεδίο εφαρμογή, πιστεύω ότι θα επιταχυνθεί η συμφωνία δεν νομίζουμε ότι θα είχε κάποια προσθέμενη αξία η δεύτερη ανάγνωση. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σχετικά κοντά στην γενική θέση του Συμβουλίου. Άρα βλέπω εδώ έναν ορίζοντα, ένα, μια ευκαιρία την οποία δεν θα πρέπει να χάσουμε. Ο πρόεδρος Χάρμπορ έκανε κάποια σχόλια. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και για να μην υπερβάλλω, ε, ίσως να μην είναι ένα ακρογωνία, ένα, ένα ορόσημο, αλλά να είναι ένα λιθαράκι. Ε, και εσείς κύριε Χάρπορ διερωτηθήκατε τι από τα δύο είναι. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μάλλον έστω και ένα λιθαράκι πάντως καλό είναι, αν είναι, για τους καταναλωτές. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί νομικοί όροι και προποθέσει στα κράτη-μέλη και νομίζω ότι ακόμη και μια πλήρης εναρμόνιση σε αυτό το στάδιο δεν θα ήταν δυνατή και εφικτή. Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι να έχουμε συμφωνία, έστω και με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Γιατί θέλουμε να αυξηθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και να ολοκληρωθεί έτσι η ενιαία αγορά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Γκέρ. Κύριος Σβάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα για το αν είναι ορόσημο ή όχι, αυτό είναι θέμα φιλοσοφικό. Πάντως για τις μεγάλες στιγμές θυμίζω τους ιδρυτές πατέρες τον Αλτιέρο Σπινέλη για παράδειγμα του οποίου το όνομα δώσαμε σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων της ομάδας μας λέει ο κ. Σφάμπα αλλά έδωσε το ΕΛΚ στην πραγματικότητα το όνομα του Αλσίτε Τεγκάσπερη λέει ο Διερμηνέας Πάντως οι τροπολογίες που οι τροπολογίες που συναποτέλεσαν συμβιβασμούς είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε. Κανένας δεν θα είναι απόλυτα ικανοποιημένος, όμως όλοι θα είναι σε θέση να ικανοποιηθούν για ορισμένα σημεία. Θα ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Ρέντινγκ για την ενθάρρυνση που μας έδωσε και απόψη στην απόψηνή συζήτηση. Ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και της Προεδρίας του Συμβουλίου. Ευχαριστώ και τον κύριο Χάρμπορ για την υπομονή που έδειξε και μαζί μου και με τους άλλους. Προς την πρώην συνάδελφο κυρία Γκέρι εκφράζω την επιθυμία να κατανοήσει και ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει ίσως να δεχθεί την κοινή θέση του Συμβουλίου όπως την ε, υιοθέτησε αυτό τους 24 Ιανουαρίου χωρίς να ζητήσει κάποιες τροποποίησεις. Ελπίζω ωστόσο αυτές να μπορέσουν να γίνουν μέσα σε ένα πνεύμα επικοδομητική συνεργασία τις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ κύριε Σβάπ. Μάλλον πρόκειται να ξενυχτήσουμε, σας προεδοποιώ. Λοιπόν, κλείνει εδώ η συζήτηση. Αύριο στι 11.30 θα ψηφίσουμε.